με την έγκριση των πρακτικών συνεδρίασής μας. Η τελευταία ανακοίνωση, η αρμόδια επιτροπή μου έχει μεταφέρει μία έκθεση σε σχέση με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα διανεμηθεί αυτή η έκθεση βάσει του άρθρου 204. Θεωρείται ότι είναι εγκεκριμένη αν τουλάχιστον αν το αργότερο 48 ε, ώρες μετά από την ε, γνωστοποίηση αυτή δεν υπάρχει μια αντίρρηση από μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 συναδέλφους για να γίνει ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Η τελική μορφή της ημέρησης διάταξης μετά από τη συνεδρία της συνέλευσης των Πρόεδρων